Παρακαλώ ησυχία, αρχίζουμε με την σημερινή μας εργασία. Θα είδατε την ημερήσια διάταξη, θα αρχίσουμε, μάλλον αρχίσαμε με τους συντονιστές. Οι εισηγητές θα μας ε, πούν τα αποτελέσματα. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια ως προς την ημερήσια διάταξη, με βάση τις, ε, τις γραπτές ενδείξεις Θα ήθελα να πληροφορήσω τους συναδέλφους και την Κομίσια ότι ο Σαλβαδόρ Γκαρίγκα αισθάνθηκε άσχημα την προηγούμενη εβδομάδα στο τέλος της Ολομέλειας. Μπήκε στο νοσοκομείο τρεις μέρες στο Στρασβούργο, τώρα είναι καλά. Και θα ήθελα, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, να του διαβιβάσω τις ευχές μας ε, για τάχιστη ίαση και ελπίζουμε να είναι μαζί μας το συντομότερο. Επίσης, ο Τζοβάνι Λαβία δεν βρίσκεται εδώ, που είναι ο εισηγητής ε, για τον προϋπολογισμό του 14, έχασε τη μητέρα του και βρίσκεται στη χώρα του για την κηδεία της μητέρας του. Εξ της Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, εκφράζω, θα εκφράσω τα συλληπιτήριά μας. Άρα τα σημεία 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης ε, αναστέλλονται και στρέφουμε προς το ΕΛΚ, το παντοδύναμο ΕΛΚ, για να πω ότι θα ήταν επιθυμητό κάποιος από την ομάδα σας να τον αντικαταστήσει για να μας μιλήσει για το σημείο 17. Ε, δηλαδή το τμήμα 3 της Επιτροπής της αιτήσει μεταφοράς πιστώσεων. Κάποιος να τον αντικαταστήσει δυνατόν. Ως προς την ημερήσια διάταξη, σας προτείνω να προσθέσουμε ένα σημείο που θα εξετάσουμε σήμερα το απόγευμα που αφορά την εξέταση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την αρμόδια αρχή για την υπογραφή του ετησίου προϋπολογισμού. Η νομική υπηρεσία και ο υπεύθυνο ο κύριος Πενέρα είναι στη διάθεση της Κομπού και σήμερα το απόγευμα θα μας ε, υποβάλει, θα μας παρουσιάσει αυτή την απόφαση η οποία ε, ικανοποιεί το Κοινοβούλιο. Οι παλαιότεροι θα θυμόσαστε αυτή τη νομική διαφορά που μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό πριν από τη συνθήκη της Ρώμης στο Συμβούλιο και φαίνεται ότι λύθηκε αυτή η διαφορά. Χρειάστηκε βεβαίως αρκετός χρόνος. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια στην ημερήσια διάταξη. Ωραία θαυμάσια. Οι άλλες ανακοινώσεις υπάρχουν στο κόμπου News. Θα ήθελα να σας πω ότι κατά τις 11 θα έχουμε μαζί μας μία ομάδα επισκεπτών του Ράιμαρ Μπέγκε, που είναι μέλη μιας οργάνωσης του κρατηδίου του, του Σλέσφι Χολστάιν. Λοιπόν, τρία. Έγκριση των πρακτικών συνεδρίασης ε, της 5ης Σεπτεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Σας προτείνω τώρα να περάσουμε στο σημείο 5, που είναι η παρουσίαση των εισηγητών μας των εισηγητριών του Γενικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 14, γνωρίζοντας ότι αν Γένσεν που συμμετέχει στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών που θα μεταβεί στο Βίλνιους, θα πρέπει να αποχωρήσει πριν από το τέλος του πρωινού, γι' αυτό θα αρχίσουμε με το δικό της θέμα. Η υπόλοιπη αντιπροσωπεία για το Βίλνιους θα αποχωρήσει λίγο αργότερα έτσι ώστε να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση μέχρι το τέλος της. Προτείνω λοιπόν στην Αν να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. The budget 2014. Ο προϋπολογισμός του 2014 είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας σε σχέση με τον προϋπολογισμό που έχει προτείνει η Επιτροπή είναι 5 με 6% πιο κάτω από τον φετινό προϋπολογισμό. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης που πρέπει να γνωρίζουμε και να καταστήσουμε σαφές προς όλους. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που ακολουθεί φθήνουσα πορεία. Και η φθήνουσα πορεία αντικατοπτρίζει την συμφωνία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου στη συμφωνία που αφορά ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο της επόμενης επταετίας. Στη συνέχεια είχαμε μερικές περικοπές από το Συμβούλιο στη δική του ανάγνωση για τον προϋπολογισμό του 2014 στις αρχές του Σεπτεμβρίου έγιναν αυτές οι περικοπές. Δεν ήταν τεράστιες σε σχέση με αυτές που γνωρίσαμε παλαιότερα. Ήταν της τάξης του 2% ως προς τις υποχρεώσεις. Και ίσως υπάρξουν νέες συμβάσεις, αλλά προς τις πληρωμές που απασχολούν τους Υπουργούς Οικονομικών, τα χρήματα δηλαδή που πρέπει να καταβάλουν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, εκεί έκαναν μία περικοπή της τάξης του 1%. Δεν φαίνεται καταστροφική, αλλά βρισκόμαστε σε δινή θέση σε σχέση με τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρώσει τους λογαριασμούς για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Και αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν θα μιλήσουμε για τον ε, προϋπολογισμό για του χρόνου στην ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Το Σαββατοκύριακο ασχολήθηκε με 1880 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στις θέσεις του Συμβουλίου οι 464 αφορούν τις επιτροπές, οι 577 από πολιτικές ομάδες και 842 από τα μεμονωμένα μέλη. Και η γενική τάση που διαγράφεται από τις εξειδικευμένες ομάδες και επιτροπές είναι ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε τον προϋπολογισμό, το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής με λίγες εξαιρέσεις, ορισμένες γραμμές όπου οι Επιτροπές είπαν ότι μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις περικοπές και υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου οι Επιτροπές και οι ομάδες κινούν πέραν αυτών των αριθμητικών στοιχείων, δηλαδή πάνω από τα στοιχεία της Επιτροπής. συζητήσαμε την κατάσταση μεταξύ πολιτικών ομάδων για να εκπονήσουμε μία στρατηγική και νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία κοινή θέση αν και υπάρχουν εκρεμή θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τις πληρωμές καταρχήν, όπου έγιναν και οι μεγαλύτερες περικοπές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ήδη φέτος αντιμετωπίζουμε ένα θέμα ότι δεν έχουν μπει αρκετά χρήματα στη γραμμή για να πληρωθούν οι λογαριασμοί του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα διαρθρωτικά ταμεία Ιδιαίτερα τα προγράμματα που ε, διέπονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή τα έργα οδοποιίας, ε, η κατασκευή ε, γεφυρών και ούτω καθεξής, αφορούν τις συμβάσεις καθεαυτές, οι οποίες υπογράφονται, αλλά μετά από χρόνια έρχονται οι λογαριασμοί προς ε, πληρωμή. Και μέσα στην επταετία πάντα βλέπετε να εισραίουν περισσότεροι λογαριασμοί και γνωρίζουμε την κατάσταση όπου οι Υπουργοί Οικονομικών, αφού έχουν υποσχεθεί στην ε, Πολωνία, στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες ή περιφέρειες, να αρχίσουν τα προγράμματα όταν φτάνουν λογαριασμοί δεν θέλουν να τους πληρώσουν και αμφισβητούν ε, τις προβλέψεις, εκτιμήσεις της Κομισιόν και υποβάλλουν ε, πολιτικά αριθμητικά, πολιτική υφή αριθμητικά στοιχεία για τις ανάγκες. Δώσαμε μεγάλη μάχη έτσι ώστε το Συμβούλιο να πληρώσει τους λογαριασμούς που είναι υποχρεωμένο να πληρώσει και είχαμε και διορθωτικούς προϋπολογισμούς τη τάξη των 11,2 δις και έχουμε 4 ε, δις, 3,9 δις που πρέπει να αποφασιστούν από το Συμβούλιο γιατί είχαμε αυτή την έλλειψη φέτος. Αυτό μπορεί να συμφωνηθεί με ειδική πλειοψηφία. Πέραν αυτού χρειάζεται ομοφωνία και ξέρουμε ότι κράτη-μέλη που ποτέ δεν θα προσυπέγραφαν. Αυτή είναι η κατάσταση φέτος λοιπόν. Τι θα γίνει του χρόνου επίσημα η Επιτροπή μας λέει ότι του χρόνου, εάν έχουν το πλήρες ποσό της οροφής του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, μπορούν να λύσουν το θέμα, γιατί θα λάβουν τα χρήματα που ζήτησαν φέτος. Όμως, ακούμε ψιθύρους στους διάφορους διαδρόμους για ελλείψεις και για ελλείμματα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με την Κομισιόν ποια είναι η πραγματική εικόνα, ποια είναι τα πραγματικά ποσά και μπορώ να πω ότι η Λιθουανική Προεδρία θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και θα διαπραγματευτούμε τον προϋπολογισμό μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας εργασίας για τις πληρωμές που θα συσταθεί για να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες για να ανταποκριθούμε στις ε, υποχρεώσεις πολλών ετών πριν. Πρέπει να πληρώσουμε τους λογαριασμούς για έργα που προαποφασίσαμε. Αυτό είναι το σωστό. Το συζητήσαμε με τους συντονιστές. Πρέπει να εκπονήσουμε μια στρατηγική <coughs> για τις ε, πληρωμές έτσι ώστε η Επιτροπή να λάβει τα χρήματα που ζητά Βεβαίως ε, θα ήταν σκόπιμο να έχουμε την πλήρη εικόνα για να πληρώσουμε όλους τους λογαριασμούς, αλλά τουλάχιστον αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε γι' αυτό και οι συντονιστές το συζήτησαν αυτό για το πώς μπορούμε να κινηθούμε πέρα από τις οροφές του σχεδίου προϋπολογισμού για τις πληρωμές και τα ποσά πάνω από την οροφή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για προγράμματα που πρέπει να ολοκληρωθούν και που χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ρευστότητα. Εδώ γίνονται συζητήσεις για το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί από τεχνικής πλευράς και κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε με το νέο έκτακτο ε, αποθεματικό 4 δις ευρώ το οποίο θα πρέπει να δούμε αργότερα. Δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το μέσο ευελιξίας. Θα τα συζητήσουμε αυτά, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί στη θέση μας διαπραγμάτευση σε σχέση με τις πληρωμές, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την, τις πληρωμές αυτές των λογαριασμών. Ως προς τις υποχρεώσεις, Έχουμε προβλήματα με όλες τις ε, τροπολογίες που εισραίουν στο κεφάλαιο 1α και 4 για τις αναπτυξιακές πολιτικές και την εξωτερική πολιτική. Βλέπουμε ότι οι επιτροπές, οι ομάδες και τα μέλη ε, επιθυμούν περισσότερα χρήματα από αυτά που ε, είχαμε σε αυτό το λιτό προϋπολογισμό, το λιτό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο συμφώνησε, επί του συμφώνησε και το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Είπαμε λοιπόν ότι θα αρκεστούμε, θα δεχτούμε τους νέους κανόνες. Είδα λοιπόν τις τροπολογίες για να δω τι μπορεί να γίνει. Στο κεφάλαιο 1, στο τμήμα 1, μας ενδιαφέρει το front loading του προγράμματος Εράσμους, το κόσμο και τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα και εκπαιδευτικά που δεν υπήρχαν στην ανάγνωση του Συμβουλίου, αλλά η Επιτροπή θα προβάλλει έναν διορθωτικό προϋπολογισμό. Θα δούμε ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Αλλά οι Επιτροπές και οι ομάδες ζήτησαν συγκεκριμένες, υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις. Όταν μιλάμε για το front loading, προσπαθήσαμε να προτρέξουμε κάπως. Άλλα προγράμματα καθυστέρησαν και ζήτησα ορισμένε ειδικέ γραμμές για την ενέργεια και το ΙΤΡΕ. Θα δούμε ποια είναι η θέση της Επιτροπής. Στο 1β δεν υπάρχουν προβλήματα. Ως προς τα διαρθρωτικά θα δείτε ε, μία κατανομή μεταξύ κρατών μελών. ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ε, κατηγορίες ε, ανθρώπων. Μερικοί θέλουν να κινηθούν πέρα από την αρχική πρόταση της Κομισιόν και υπάρχει και το θέμα του front loading της πρωτοβουλίας για τους νέους και αυτό είναι το βασικό θέμα στο 1β σε σχέση με τη γεωργική πολιτική δεν έχουμε προβλήματα. Η Επιτροπή Γεωργίας σε σχέση ε, με το, το φαγητό στα σχολεία και τα φρούτα στα σχολεία ε, ζητά επιπρόσθετα κονδύλια. Αυτό το τμήμα δεν αποτελεί ε, πρόβλημα και για το τμήμα 3-2 έχουμε αυξήσει τα ποσά σε σχέση με την αρχική πρόταση του Συμβουλίου για πολιτισμικά προγράμματα για τα προγράμματα, προγράμματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, προγράμματα υγείας και υπάρχουν ορισμένοι οργανισμοί σε αυτόν τον τομέα. Ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες σε σχέση με την υγεία και μετά στον, ε, στο προσχέδιο προϋπολογισμού κινούμαστε λίγο πέραν από τα αρχικά ποσά, ιδιαίτερα για τους ε, οργανισμούς που έχουν νέα καθήκοντα και χρειάζονται τα σχετικά κονδύλια για να ανταποκριθούν. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι στο, το τμήμα 3 δεν θα αποτελέσει πρόβλημα. Μετά όμως έχουμε την ε, πολιτική την εξωτερική πολιτική και εδώ έχουμε μεγάλα προβλήματα για να ανταποκριθούμε στα, στις επιθυμίες μας. Η Επιτροπή Ανάπτυξης θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουμε τον ίδιο προϋπολογισμό για τα φτωχά κράτη-μέλη ε, και του χρόνου όπως και φέτος. Και ως προς το DMFF, αυτό που προβλέπετε είναι μεγάλες περικοπές. To go back to the uh, commission's figures. Αυτό προβλέπετε στις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Και η Επιτροπή Απασχόλησης εξέφρασε την επιθυμία της να αλλάξουμε την διάρθρωση ορισμένων γραμμών του προπολογισμού για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για το πώς δαπανώνται τα, τα κονδύλια. Η ΑΦΕΤ ζήτησε περισσότερα κονδύλια από αυτά που προβλέπονται στην οροφή. Προσπαθούμε να λάβουμε περισσότερα χρήματα και εδώ οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες ήταν πιο μετριοπαθής από την ε, Επιτροπή ΑΦΕΤ. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να βρούμε μια κοινή λύση. Οριακό θα είναι το κατά πόσο θα βρεθούμε πάνω ή κάτω από την οροφή. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που θεωρούν ότι πρέπει να κινηθούμε πέραν της οροφής και να χρησιμοποιήσουμε τα ευέλικτα μέσα το μέσο ευελιξίας. Στην αρχική μας πρόταση θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο ευελιξίας για ένα μικρό ποσό, για μία αύξηση στα ποσά για την Παλαιστίνη, γιατί θα πρέπει να γίνει μία αύξηση γιατί ίσως και το ελεγκτικό συνέδριο στην ε, έκθεσή του εκφράσει επικρίσεις για την διαχείριση των ταμείων. Γι' αυτό θα θέλαμε η Επιτροπή να μας απαντήσει τάχιστα πριν ζητήσουμε περισσότερα χρήματα. Αυτά για την κατηγορία 4. Ε, η Επιτροπή, οι Επιτροπές ντεβεκε. και ΑΦΕΤ εξέφρασαν λοιπόν αυτές τις επιθυμίες και προσπάθησα να ανταποκριθώ σε αυτές τις προτεραιότητες των δύο επιτροπών. Μετά υπάρχουν τα διοικητικά έξοδα. Θα έλεγα ότι οι βασικές ε, εξηγήσει θα πρέπει να προέλθουν από την κυρία Χόλμαϊρ, θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση όταν μιλάμε για άλλα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ασφαλώς η μεγάλη δυσκολία εδώ θα είναι η υπόθεση, η δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί ακόμα για τις, ε, τους μισθούς. Η πρώτη άποψη που παρουσίασε το δικαστήριο είναι ότι θα χάσει το δικαστήριο και ότι θα πρέπει πολύ απλά να πληρώσουν τα χρήματα. Αλλά φυσικά αυτό είναι δύσκολο εάν δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω γενικά σε ό,τι αφορά τις ε, υπηρεσίες, τους οργανισμούς. Βλέπουμε ότι αρχικά υπάρχει, υπήρχε η στρατηγική σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες αυτές τις ε, αποκεντρωμένες. Συμφωνήθηκε περικοπή 5% συμφωνήσαμε κι εμείς ε, σε ό,τι αφορά τις περικοπές αυτές, σκεπτόμενοι ότι θα παρατείνουμε το ωράριο εργασία. Και άρα θα χρειαζόμαστε θεωρητικά λιγότερο προσωπικό. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι στο μέλλον η ανάπτυξη κάποιων υπηρεσιών θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από μειώσεις σε άλλες υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς αυτούς. Ε, πρόκειται για λειτουργικές δαπάνες των οργανισμών αυτών. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τέτοιες περικοπές και τέτοιες ε, οικονομίες κλίμακας, ε, για παράδειγμα μέσω ε, συγχώνευσης οργανισμών. Είναι ανοιχτή η Επιτροπή Προϋπολογισμών σε τέτοια ενδεχόμενη λύση, αλλά το Συμβούλιο φαίνεται ότι αντιστέκεται, γιατί θέλει ο καθένα να κρατήσει το δικό του οργανισμό στο, στην κάθε χώρα. Άρα θα πρέπει να εξεταστεί η αξία κάθε οργανισμού ξεχωριστά και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του και σε ό,τι αφορά τις περικοπές των δαπανών. Κάτι που συμπεριέλαβα ήταν ένα σημείο το οποίο επέβαλε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ζήτησε πιο πολλά κονδύλια λόγω της αύξησης των αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά τις ρυθμιστικούς οργανισμούς στον τομέα των ε, ε, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και περικόπηκαν κάποιες γραμμές και έτσι βρήκαμε νέα κονδύλια. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι σωστός τρόπος αντιμετώπισης, να βρίσκουμε τα κονδύλια από περικοπές σε άλλες ε, γραμμές. Συμπεριλαμβάνουμε λοιπόν την πρόταση τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων σε ό,τι αφορά τα πολιτικά project και τι προπαρασκευαστικέ δράσει. Πολλέ είναι οι επιθυμίε που ακούστηκαν από κράτη-μέλη, από τι επιτροπέ, από του βουλευτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την άποψη επί των προτάσεων αυτών, την τοποθέτησή τη. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερω. Είναι πολύ ωφέλιμο αυτό το υλικό για το έργο μας. Επίσης, διευκρινίσαμε ότι ενδεχομένω να μην χρησιμοποιήσουμε μόνο τη γραμμή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένως, αλλά οι πληροφορίες αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες και ωφέλιμες για μας κατά τη λήψη αποφάσεων. Πολλά από αυτά τα πολιτικά προγράμματα για τις δράσεις έχουν λάβει έμφαση γιατί καλύπτονται από ήδη υφιστάμενα προγράμματα. Άρα περνάμε σε επίπεδο λεπτομεριών. Δεν έχουμε ακόμα διευκρινίσει τις λεπτομέρειες αυτές, αλλά βρίσκομαι σε φάση διαπραγμάτευση με τις πολιτικές ομάδες για να καταλήξουμε σε ένα πακέτο πληθυκών προγραμμάτων, προπαρασκευαστικών δράσεων, για να μείνουμε εντός των ορίων στο πακέτο αυτά και φυσικά να τηρήσουμε και τα όρια, τα ανώτατα των διάφορων ε, τίτλων. σε θέματα διαφάνειας σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που χορηγούνται στα κράτη-μέλη για να διαχειριστούν την φόρο συλλογή και άλλων ίδιων πόρων. Εδώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε διαφάνεια και καταλαβαίνω ότι ο Πρόεδρός μας θα δράξει την ευκαιρία για να γίνει μια τέτοια συζήτηση στην Επιτροπή στο θέμα, για το θέμα των ίδιων πόρων. Η αλλαγή των γραμμών δεν, ε, σε ό,τι αφορά τους πόρους δεν αλλάζει την ε, γραμμή των δαπανών, των πόρων. Είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Και μετά έχουμε και το θέμα, πέρα από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης, το απόθεμα αυτό. Νομίζω ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και θα πρέπει να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε του χρόνου για τη Συρία. Όπου ενδεχομένω οι ανάγκε να είναι τεράστιες. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το σκεφτούμε. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές της στρατηγικής την οποία εξετάζουμε. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η στρατηγική θα πρέπει να είναι πολύ δυναμική σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Αυτό δεν το κάναμε παλαιότερα γιατί δεν ήταν προβληματικό. Τώρα όμως πλέον έχει καταστεί πρόβλημα. Το Συμβούλιο δεν προτίθεται. να δώσει στην Επιτροπή αυτά που χρειάζεται για να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Δηλαδή προτείνεται μια συγκεκριμένη στρατηγική με πολύ σαφείς στόχους. Έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή ε, για τον προπολογισμό αν ε, τα ξέρω καλά το Σώμα των Επιτρόπων σήμερα ε, θα αποφασίσει το ιδιορθωτική επιστολή... ή όχι... <laughs> κύριε Διευθυντά ναι όντως η επιστολή αυτή θα φτιαχτεί την επόμενη εβδομάδα αλλά Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει μια διόρθωση στο διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 6 σχετικά με τους πόρους. Θα θυμάστε ότι σε αυτόν τον προϋπολογισμό είχαν μειωθεί τα έσοδα ε, στον τίτλο των ε, παραδοσιακών ε, ίδιων πόρων και τα έσοδα από τα πρόστιμα ε, είχαν μειωθεί οπότε οι εισφορές ως ε, με τη μορφή του RNB θα έπρεπε να αυξηθούν και ε, υπάρχουν ε, ε, και άλλες δαπάνες ε, υπάρχουν ε, υπάρχει επίσης όσο και παράξενο σας φαίνεται των μέσων δασμών τελωνιακών δασμών γιατί, γιατί έχουμε κρίση ουσιαστικά στις εισαγωγές Λοιπόν, αυτός ο διορθωτικός τους προϋπολογισμός επαριθμών 6 πρέπει να διορθωθεί ξανά διότι δυστυχώς πραγματικά επιβεβαιώθηκε και αυτή η μείωση των εσόδων από τους τελωνιακούς δασμούς πρέπει λοιπόν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι εισφορές RNB ένα δις 400 εκατομμύρια περίπου είναι το κενό που πρέπει να καλύψουμε τα πρόστιμα είναι 600 εκατομμύρια περίπου Αυτά λοιπόν θα τα πει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τα αποφασίσει και για να συμπληρώσει την ολικόνα για το... Αυτά για να συμπληρωθεί η εικόνα για το 2013 και την επόμενη εβδομάδα έχουμε την πρώτη διορθωτική επιστολή για το προεπολογισμό του 2014. Λαμασούρ, ωραία, ναι, αλλά έχουμε και τη δεύτερη δόση του DAB δηλαδή 3,9 ναι ναι η Επιτροπή θα αποφασίσει τον προϋπολογισμό τον διορθωτικό υπαριθμών 8 που υπάρχει το DAB 2α και έχουμε και τα γεωργικά λέει ο κ. Λαμασούρ βεβαίως παρακαλώ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί η συγγήτρια μας περιέγραψε αρκετά λεπτομερώς το πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Σήμερα το πρωί ακούσαμε μια αντίστοιχη παρουσίαση και έγινε και άλλη μια συζήτηση για την ενδεχόμενη στρατηγική του Κοινοβουλίου. Οι περισσότερες προτάσεις των σοσιαλιστών ελήφθησαν υπόψη από τη, στην τελευταία πρόταση της εισηγητρίας και, αλλά υπάρχει και κάτι τι άλλο που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. 6% τα μείωση υπάρχει στον προπολογισμό του 2014 σε σχέση με το προϋπολογισμό του 2013 και αυτές οι μειώσεις θα πρέπει να καλυφθούν από κονδύλια από προγράμματα που όμως ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους σοσιαλιστές παραδείγματο χάνει δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη κτλ και συνεργασία για την ανάπτυξη πάντα τα ποσά για την ανάπτυξη ήταν χαμηλότερα από ό,τι ε, φανταζόμαστε και από ό,τι θα έπρεπε να διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παίκτη στο θέμα αυτό λοιπόν η κυρία Γένσεν βέβαια ο, επαναλαμβάνω δέχθηκε για τις υποχρεώσεις τις περισσότερες ε, προτάσεις μας. Αλλά για τις πληρωμές τώρα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση σε αυτή την Επιτροπή για να ορίσουμε τη στρατηγική και το πώς θα προχωρήσουμε τι θα, θέση θα κρατήσουμε στις ε, επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Η πρόταση των σοσιαλιστών ήταν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε και το ολόκληρο το περιθώριο που έχουμε για τα, αυτό που ονομάζουμε contingency margin, τα τέσσερα δις δηλαδή. Γιατί λέμε ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σχεδόν ολόκληρο αυτό το απόθεμα δεν ξέρω, ίσως αυτό επιβεβαιωθεί και την επόμενη εβδομάδα από τον τριμερή διάλογο, αλλά γιατί εμείς πιστεύουμε ότι θα καταλήξουμε να έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης των 12 δις για φέτος. Δεν υπάρχουν νούμερα, αλλά υπάρχουν και φήμες που μιλάνε για 20 δις έλλειμμα. Λοιπόν, το μέσο αυτό το οποίο ουσιαστικά α, ουσιαστικά για τις πληρωμές αλλά είναι για τις υποχρεώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις πληρωμές διότι όταν μιλάμε για διψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων δεν μπορούμε να καλύψουμε πουθενά άλλου αυτό το ποσό εκείνο που πιστεύουμε όπως το είπαμε, το λέμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι ότι σίγουρα έχουμε πρόβλημα στις πληρωμές η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις και δεν μπορούμε να δεχόμαστε να υπάρχουν ελλείμματα και κενά στις πληρωμές και όχι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση και οι περιφέρειες αλλά και τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις, ιδιωτικές, ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να αντέξει να μην επιστρέφονται τα χρήματα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά όμως δεν ξέρω πού θα τα βρούμε τα 12, τα 20 δις. Νομίζω ότι αυτό το ποσό θα μπορούσε να συμφωνηθεί, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Χρειαζόμαστε 20 δις. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, τη στιγμή που μπορούμε να ζητήσουμε 4 δις, γιατί να μην το κάνουμε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Υπάρχει ένα προσχέδιο συμβιβασμού το οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Για τις πληρωμές θα πρέπει να συμφωνήσουμε για την στρατηγική του Κοινοβουλίου και ποια θα είναι η στάση μας προς το Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει το Συμβούλιο δεν θέλει να δώσει τα χρήματα, αλλά το Κοινοβούλιο δεν ε, μπορεί να το δεχτεί αυτό. Δηλαδή είναι ε, ε, υποχρεωτικό, πρέπει να πληρωθούν οι λογαριασμοί. Πώς να το κάνουμε. Και φαίνεται ότι στο Συμβούλιο ανέκυψε από μία χώρα το θέμα της καταβολής των λογαριασμών. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να επιμείνει για να πληρωθούν οι λογαριασμοί. Θα δούμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα κατά πόσο θα έχουμε πιο επίσημα στοιχεία από την Επιτροπή και το Συμβούλιο και να αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση μιας ανωδικής πορείας, διότι δεν είναι θέμα του Κοινοβουλίου. Πρέπει να πληρωθούν οι λογαριασμοί γιατί οι χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλες ε, δυσκολίες και υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα. Ε, χώρες ε, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πληρωμές είναι αυτές τις οποίες χρωστάμε περισσότερα χρήματα. Δηλαδή επιδεινώνεται η κατάσταση και το Συμβούλιο θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούμε να, να χρωστάμε 20 δις στα κράτη στα κράτη, στις επιχειρήσεις, στις περιφέρειες και να μην τα καταβάλουμε. Θα πρέπει να φτάσουμε λοιπόν σε μια συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σαρτόγκ. Eh, Σας ευχαριστώ συνάδελφε για την σύνοψη αυτή. Δύο σημειώσεις έχω να κάνω τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι κάνουν απάτες όλο και πιο πολύ με τα δραστηριοτικά ταμεία και θα χρειαστεί λοιπόν μεγαλύτερο έλεγχο από τι δύο επιτροπέ του Κοινοβουλίου και το Ελεκτικό Συνέδριο ε, Ετησίω ελέγχει για τα σταλίε, αλλά ο κύριο Φαν δεν συμφωνεί γιατί θέλει να κάνουμε θετική διαφήμιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σημειώσω ότι με ικανοποιεί ωστόσο το έργο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θεωρώ ότι καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί εκ των προτέρων παρά να προσπαθούμε εκ των υστέρων να διορθώνουμε τα, τις αντασταλίες. σε ό,τι αφορά τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου πολλές δαπάνες διαγράφονται σε διάφορα περιφερειακά και ταμεία νομίζω ότι καλύτερα να είμαστε όπως σας είπα εκ των προτέρων πιο προσεκτικοί και πιο προληπτικοί παρά να λυπούμαστε εκ των υστέρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καλύτερη διαφάνεια, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. Μιλάτε για αυτή εσείς, όμως και ο συνάδελφός σας, ε, Μούλερ, κάνετε μια τροπολογία για να διαγραφεί αυτή, να μειωθεί αυτή η διαφάνεια. Τι να πω, εγώ το βρίσκω πραγματικά παράδειγμα αυτό. Ευχαριστώ. Merci, mon cher. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Ζητεί το λόγο Ιάν Γέννησεν για να κλείσουμε το θέμα. Όχι, για να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτό το διορθωτικό προϋπολογισμό και αυτό το περίφημο front loading, την κατά ε, αντιμετώπιση κάποιων προγραμμάτων. Δηλαδή η έρευνα, το Εράσμος και το Κόσμι έχουν υψηλή προτεραιότητα. Oui, ce que nous a dit, monsieur. Ναι, λέει ο πρόεδρος, αυτό που είπε ο κύριος Ζωνζόν και ας με διορθώσει αν κάνω λάθος μας είπε λοιπόν ότι η διορθωτική επιστολή που θα ασχοληθεί ακριβώς που θα καλύπτει και αυτό το front loading δηλαδή όλα αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία εισήχθησαν μέσω του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου η επιστολή αυτή θα αποφασιστεί την επόμενη εβδομάδα μαζί με τη δεύτερη δόση των πληρωμών του, ε, του προϋπολογισμού 2013. Θα είναι ο διορθωτικός προϋπολογισμός υπαριθμών 8. Λοιπόν, προχωρούμε. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια-δυο ερωτήσει έχω. Θα ήθελα να θέσω. Πρώτα-πρώτα η Αν Γέννησεν είπε ότι εσείς Μπορεί να έχετε κάποιες καινούργιες ιδέες για τους ίδιους πόρους. Εγώ λέω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τους ίδιους πόρους. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα γιατί δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο. Αν πρέπει να σεβαστούμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και υπάρχει βέβαια και η ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με αυτό αλλά θα ήθελα να με διαφωτίσετε για τις καινούργιες ιδέες που ενδεχομένως να υπάρχουν. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα πρώτα για την ε, δικαστική υπόθεση για τους μισθούς. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι αριθμοί, ε, μιλάμε μόνο για εκκρεμούσες αυξήσεις του 11 ή προχωρούμε και παραπάνω κάτω θα πρέπει να πληρωθούν αυτές το 13 ή το 14 αν έχουμε περισσότερο περιθώριο γιατί αν πρέπει να κάνουμε τις πληρωμές αυτές το 13 είναι τεράστιο το βάρος και για το κομμάτι του προπολογισμού που αφορά στην Κομισιόν αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως ε, προσπαθούμε ε, με νύχια και με δόντια να, κατέβ, να φτάσουμε στο επίπεδο του πληθωρισμού άμα έχουμε να πληρώσουμε και τις αυξήσεις στους μισθούς καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αφόρητα. Τέλος, ξέρουμε τίποτε παραπάνω για το πόσο θα κοστίσουν οι απλήρωτοι λογαριασμοί γιατί ήδη βρισκόμαστε πληρώνουμε υπερβολικά αργά και το να πληρώνουμε αργότερα από ό,τι πρέπει να πληρώνουμε πόσο μας κοστίζει αυτή είναι η ερώτηση είναι, από πολιτική άποψη είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι τι μας κοστίζει η ε, πληρωμή των λογαριασμών μας αργότερα από ό,τι θα έπρεπε ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος να απαντήσω αμέσως ε, για τους ίδιους πόρους υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία όμως αλληλοσυμπληρώνονται δηλαδή ε, βοηθούν για την επίτευξη του ίδιου στόχου πρώτον αυτή τη στιγμή κάνουμε ανταλλαγή από, έχουμε ανταλλαγή απόψε μεταξύ των τριών οργάνων για τη δημιουργία μιας ε, ομάδας υψηλού επίπεδου που θα ασχοληθεί με τη μεταρρύθμιση των ε, δημοσιονομικών της Ένωσης. Προβλέπεται αυτό από το πολυονομικό, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και λέγεται εκεί ότι τώρα το φθινόπωρο θα φτιαχτεί η ομάδα αυτή, θα οριστούν από τα τρία όργανα τα μέλη της ομάδας αυτής και αυτή τη στιγμή εμείς ανταλλάζουμε απόψεις για τον αριθμό των μελών, για τη σύνθεση, για το θεματολόγιο και για το χρονοπρόγραμμα εργασίας. Ε, έχουμε την επίσκεψη στο Βίλνιους αύριο και εκεί θα συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Ριμποσκάιτε, την πρόεδρο της Λιθουανίας που γνωρίζει βεβαίω τα του προπολογισμού. και στα πλαίσια της ομάδας επαφής που προεδρεύει ο Σούλτς θα πάρθει η τελική απόφαση. Θα τα πούμε με τους συντονιστές μέχρι τότε. Παράλληλα με αυτό και για να εντείνουμε την πολιτική πίεση για την σύσταση και τη λειτουργία αυτής της ομάδας για τους ίδιους πόρους πρότεινα εγώ φέτος για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια να γίνει μια συζήτηση για το σκέλος των εσόδων του προπολογισμού. Ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι για τα έσοδα οι νομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου είναι ισχνές. η δουλειά που κάναμε στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου οι διαπραγματεύσεις που είχαμε γι' αυτό το πλαίσιο για τα ή τους ίδιους πόρους μας οδήγησαν στο να πιστέψουμε ότι αν θέλουμε να υπάρχει μια ελάχιστη στήριξη από τις κυβερνήσεις ή τουλάχιστον από κάποιες κυβερνήσεις, από τα μίντια, από τους πολίτες θα πρέπει να δώσουμε πληροφορίες που δεν δίνονταν μέχρι τώρα λόγω χάρη. να πούμε ότι πρακτικά το σύστημα GNI είναι ένας φθήνων φόρος έτσι και η, όσο πιο μεγάλες είναι οι χώρες τόσο πιο πολύ συνεισ... όσο πιο μεγάλες χώρες τόσο λιγότερο συν, ε, συνεισφέρουν, μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ τους συνεισφέρουν. Όσο πιο φτωχές χώρες τόσο περισσότερο συνεισφέρουν αναλογικά να το πούμε αυτό, να φτιάξουμε ένα πίνακα, να οργανώσουμε μια συζήτηση, να αρχίσει να ενδιαφέρεται ο πολίτης για, το, ε, για τα πράγματα αυτά. Ίσως θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πιο μπροστά, αλλά το σκεφτήκαμε αυτό όταν συνειδητοποίησαμε ότι έχει τέρα είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε κάποιες ε, κυβερνήσεις να αλλάξουν το σύστημα αυτό το οποίο ουσιαστικά ήταν ε, εξ αρχής θνησιγενές αλλά τέλος πάντων λοιπόν από εκεί και πέρα έχουμε τον τους τον συνάδελφο τον Κάλβιν ο οποίος μαζί με τον Τεάννα είναι οι συγητές για τον προπολογισμό, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 14-20 ε, 2014-2020 θα τα κουβεντιάσουμε τα πράγματα αλλά ε, θα καταλαβαίνετε ότι αυτά που λέω ουσιαστικά έχουν ε, και μια παιδευτική αν θέλετε δεν ε, θέλουμε απλώς να περιπλέξουμε τις διαπραγματεύσεις προσθέτοντας κάποιες παραμέτρους. Ε, ε, θα τα δουν τέλος πάντων οι ε, συντονιστές. Θα δούμε. Λοιπόν, Χέλγα και μετά θα ζητήσω από το Γενικό Διευθυντή να απαντήσει την την ερώτηση του Κοράν που αφορούσε την Κομισιόν. Η γενική κατάσταση είναι αυτή που παρουσίασαν πολλοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε και την Άννα για την παρουσίαση. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση. Ε, βλέπουμε ότι περιορίζεται, περικόπτεται ο προπολογισμό. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μεγάλη μείωση για πρώτη φορά. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου κανονικά θα χρειαζόμασταν πιο πολλού πορού και αντιμετωπίζουμε μια... και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έχει την τόλμη να κάνει αυτά που χρειάζονται. Να σας πω τώρα ότι εμείς ε, θεωρούμε ότι καλό είναι να απορροφηθεί ε, όλο το περιθώριο που υπάρχει ε, αλλά σε ό,τι αφορά το περιθώριο για προβλεπτές ανάγκες έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Είναι ένα ε, έκτακτο μέσο, άρα front-loading, αρχική επιβάρυνση εκ εξορισμού. Δεν είναι λύση λοιπόν για το επίπεδο πληρωμών. Θα προτιμούσαμε να πιέσουμε το Συμβουλίο και να τροποποιήσουμε τον προπολογισμό και να αλλάξει το επίπεδο των πολιτεών δημοσιονομικών προοπτικών. Γιατί δεν έχει νόημα να μεταθέσουμε το πρόβλημα κάποια χρόνια για επίπεδο δεσμεύσεων, για το επίπεδο δεσμεύσεων για την επικεφαλίδα 1α και 4 έχουμε θέμα. Και δεν μας ε, ικανοποιεί μόνο το front loading. Θέλουμε αύξηση του, του ορίζοντα του κόσμου και του ράσμους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ευρυζωνικά προγράμματα έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει αναλογικότητα. Θέλουμε άλλη κατανομή. Επίσης θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τα περιθώρια και πιο πολύ ευελιξία ως τώρα χρησιμοποιείται το Flex 172 προς το παρόν και αυτό θεωρούμε ότι δεν επαρκεί. Να σας δώσουμε τώρα κάποια ιδέα τι γίνεται στις άλλες γραμμές. Επικεφαλίδα 1 Β. Εδώ είμαστε υπέρ της αύξησης ε, της βοήθειας προς τους ε, στα άτομα που έχουν ανάγκη, αλλά σε ό,τι αφορά την απασχόληση των νέων λόγω εφαρμογής θα θέλαμε να κοιτάξουμε τις δεσμεύσεις. Στην επικεφαλίδα 2 θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια θέματα εσωτερικά, αλλά θέλουμε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Ε, στην επικεφαλίδα 3, εντάξει, υποστηρίζουμε, έχουμε κάποια προβλήματα με το Frontex. Το 4 έχουμε μεγάλα προβλήματα, όπως είπατε και εσείς. Ιδιαιτέλος, μας ενδιαφέρει Το μέσο ευελιξίας για τις γραμμές DCI. Και πάλι έχουμε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τις περικοπές των μισθών. Γιατί είναι θέμα, όπως είπατε, σημαντικό ε, για τους οργανισμούς Frontex, όπως είπατε και εσείς, από πλευράς εσόδων τώρα. Νομίζω ότι καλό θα είναι να περιληφθούν στον προπολογισμό του πιο πολύ τα πρόστιμα και νομίζω ότι πραγματικά θα κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια εκεί πέρα. Ευχαριστούμε. Ο Ντομινίκ Ρικέ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω τη θέση μας ως προς την κατάσταση του προϋπολογισμού, ως προς τις πληρωμές στις οποίες προναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες, ή εξέφρασε πολύ καλά την ε, κατάσταση. Όμως δεν ε, δεχόμαστε ε, τις ίδιες λύσεις. Η θέση του ΕΛΚ είναι ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι την οροφή και να αφήσουμε το μέσο ευελιξίας καθώς και το έκτακτο περιθώριο. Γιατί να μην ε, τα χρησιμοποιήσουμε σε σχέση με την κατάσταση, διότι το πρόβλημα που ανακύπτει συνέχεια σχετίζεται με ένα επίπεδο το οποίο είναι ε, πάνω από το μέσο ευελιξίας και το, αποθεμα, το έκτακτο αποθεματικό. Υπάρχει όμως και ε, ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί το οποίο έθιξαν και οι πράσινη. Δηλαδή, εμείς χρησιμοποιούμε τα δικά μας χρήματα για τις ε, πληρωμές. Εάν χρησιμοποιούμε το ε, μέσο ευελιξίας ή το έκτακτο αποθεματικό, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε μια σχετική συμφωνία. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε εάν ε, μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε το γενικό θέμα των πληρωμών ή να χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας μέσα για να δούμε κατά πόσο ε, υπάρχει επάρκεια. Γι' αυτό η θέση του ΕΛΚ είναι ε, λογική, δηλαδή δεν θέλουμε να πάμε πέρα από τα περιθώρια ως προς το μέσο ευελιξίας και το έκτακτο αποθεματικό είναι πολύ κακή εικόνα που προβάλλουμε προεκλογικά και από πλευράς ε, ποσών ή μέσου δεν έχει νόημα να ε, καλύπτουμε με τα δικά μας μέσα τα ασφάλματα του Συμβουλίου. Ο, αντίθετα, ως προς τις υποχρεώσεις, νομίζω ότι υπάρχει βάση συμφωνίας μεταξύ των ομάδων. Αν δεχόμαστε και μία συζήτηση για το backloading, όμως δεν δεχόμαστε την πρόταση της εισηγήτριας για τα δίκτυα επικοινωνίας και την ανάπτυξή τους που δεν είναι προτεραιότητα του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια. Και σε σχέση ε, με τα ε, διαρθρωτικά ταμεία θεωρούμε ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να μετατραπεί σε μια πραγματικότητα, δημοσιονομική ε, πραγματικότητα, ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων. Στον τομέα 2 δεν θέλουμε οι άμεσες ε, πληρωμές να περάσουν στις υποχρεώσεις στο δεύτερο πυλώνα. Οι άμεσες πληρωμές είναι πολύ σημαντικές στον αγροτικό τομέα. Θα πρέπει να δούμε τι θα αποφανθεί η σχετική επιτροπή. Στον τομέα 3 δεν έχουμε σχόλια και στον 4, στο τμήμα 4 δεχόμαστε αυτό που ελέγχθη ότι υπάρχει στρέβλωση της πρότασης της Επιτροπής σε σχέση με την τελική πρόταση του Συμβουλίου και των ορμοδίων Επιτροπών, γιατί βρισκόμαστε πέρα από το περιθώριο, δηλαδή κάτω από αυτό που αρχικά ε, προτάθη. Ακόμα και στο απόθεμα τα 50 εκατομμύρια για την Παλαιστίνη, γιατί γνωρίζουμε την εισήγηση του ελεγκτικού συνεδρίου, αφορούν μια πολιτική συζήτηση του Κοινοβουλίου. Άρα σημεριζόμαστε τις ανισχύες και τις αναλύσεις της εισηγήτριας. Οι θέσεις μας για τις πληρωμές είναι ε, λίγο διαφορετικές γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα μέσω του 2014 κατά των μέσων που διαθέτουμε. Ως προς τις υποχρεώσεις το θέμα θα είναι πιο εύκολο. Μπορούμε να δεχτούμε τη θέση της εισηγήτριας και των αρμοδίων επιτροπών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ναράγχο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εντάχει θα ήθελα να σχολιάσω ε, καταρχήν ευχαριστώντας την εξαιρετική εργασία της συναδέλφου και δέχομαι αυτά που είπε ο κύριος Ρίκε Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Ποια στρατηγική θα ασχοληθούμε, για, θα, ε, ποια στρατηγική θα μας απασχολήσει για να ανταποκριθούμε στις πληρωμές και τις υποχρεώσεις. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει σαφήνεια, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι εκρεμείς λογαριασμοί, γιατί δεν μπορούμε να προβάλλουμε μια στρατηγική τη στιγμή που υπάρχουν ε, πολλές ε, διακλαδώσεις. χωρίς να έχουμε σαφείς ε, πληροφορίες και διαφάνεια. Και αυτό αφορά όχι μόνο τους βουλευτές αλλά και τους πολίτες. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Όπως είπε και ο πρόεδρος, Τη στιγμή που πρόκειται για μία παιδαγωγική άσκηση για τους πόρους μας. Πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών μας και έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τι σημαίνει προϋπορογισμός της Ένωσης. Ε, εάν λοιπόν δεν αναμορφωθεί το σύστημα θα ακολουθήσουμε την οδό που γνωρίζουμε, αλλά θα πρέπει και από παιδαγωγικής καθαρά πλευράς να πούμε και να εξηγήσουμε πώς φτάνουμε σε αυτούς τους πόρους. Γι' αυτό χρειάζεται ένας ανοιχτός διάλογος για να έχουμε σαφή θέση και να μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτείται διαφορετικά και το Κοινοβούλιο έχει άλλες αρμοδιότητες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Γιατί δεν μπορούμε να εξηγήσουμε σε έναν πολίτη πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στην ανταπόκριση ε, στις ανάγκες για αυτούς τους πόρους. Ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο πώς ε, φτάνουμε στη διαμόρφωση του ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να φτάσουμε στη ρίζα της ε, κακοδαιμονίας, να θέσουμε το θέμα από τα κάτω προς τα πάνω και για τις ε, πληρωμές χρειάζεται διαφάνεια. Το είπα, χρειάζονται γνώσεις και για να έχουμε οποιοδήποτε στοιχείο στρατηγικής θα πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Όπως σας είπα, έχουμε την επίσκεψη μίας αντιπροσωπής από το Σλέσβι Χολστάιν, ε, προσκεκλημένη του Ράιμαρ Μπέγκε, ε, να καλωσορίσουμε τους φίλους από το Σλέσβι Χολστάιν. Ε, προσέρχεστε μία στιγμή που έχουμε την πιο σημαντική συζήτηση του έτους για το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014 πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα, ποιες είναι προτεραιότητες, πώς γίνονται, πώς γίνονται οι χρηματοδοτήσεις και ούτω καθεξής. Ε, χαιρόμαστε για την παρουσία σας. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, θέλετε να απαντήσετε. Έχετε το λόγο για τα ερωτήματα των συναδέλφων. Για, ως προς τον Γκέραν Φέρμ, για τις καθυστερήσεις των πληρωμών. δώσαμε προτεραιότητα στις ε, πληρωμές προς δικαιούχους όπου εάν δεν καταβάλλονταν τα χρήματα θα έπρεπε να καταβληθούν τόκοι περιμερίας. Δηλαδή υπήρξε αυτή η προτεραιότητα. Δηλαδή ως προς τα κράτη για να μην καταβληθούν αυτοί οι τόκοι περιμερίας. Άρα δεν υπάρχει ένα, για να μην υπάρχει ένα επιπρόσθετο ε, κόστος ε, από τις ε, πληρωμές για δικαιούχους οι οποίοι προστατεύονται σε περίπτωση ε, καθυστέρησης, δηλαδή καταβάλλονται αυτοί οι τόκοι περιμερίας. Ως προς τις προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας ε, του Δικαστηρίου θα αποφανθεί για το 2011. Το Δικαστήριο θα αποφανθεί, θα τελεσιδικήσει η απόφασή του μέσα σε τρεις με έξι μήνες. Από όσο γνωρίζουμε, μέχρι το τέλος του έτους. Αλλά θα αποφανθεί για το 2011 και Αν τώρα το δικαστήριο ακολουθήσει τη θέση του Γενικού Ισαγγελέ και αν υπάρξει ανάκτηση χρημάτων, όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες να κάνουν τις ε, μεγαλύτερες καταβολές για το 2013 αυτό μπορούμε να το προωθήσουμε με βάση τη συμφωνία για το πάγωμα των μισθών, όπως, προβλέπουν, ε, όπως προβλέπει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό αφορά το 13 και πρόκειται, έχει η απόφαση αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο, άρα θα γίνει πάγωμα μισθών και δεν θα αναπροσαρμοστούν στο τέλος του έτους. Αλλά αυτό δεν επαρκεί. Θα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους χρηματοδότησης και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν την κατάσταση για να βρουν πηγές χρηματοδότησης. Ως προς την ερώτηση, το ερώτημα του κυρίου Ναράνχο για τις, ε, τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν, θα ήθελα να πω τα εξής. Οι εκτιμήσεις μας βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους οικονομικούς φορείς και ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη. Ως προς, τους, προς τα ταμεία που υπάρχει κοινή διαχείριση δεύτερον. Όσον αφορά τις πληρωμές που είναι υποχρεωτικές μέχρι το τέλος του έτους, η εκτίμησή μας είναι ότι με τα 11,2 δις θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα ποια θα είναι τα ποσά στο τέλος του έτους. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο προς το τέλος του έτους Υπάρχουν ε, σοβαρά αιτήματα καταβολής πληρωμών. Έχουμε ορισμένες ενδείξεις για τις προθέσεις των κρατών μελών μέχρι το τέλος του έτους, αλλά αυτές οι ενδείξεις είναι σχετικές. Πέρσι συζητήσαμε τις εκτιμήσεις των κρατών μελών που μας έδωσαν ένα χι αριθμητικό στοιχείο με μια συγκεκριμένη διάρθρωση και μετά είχαμε ένα άλλο ποσό το οποίο υπερεύαινε το αρχικό αλλά με διαφορετική διάρθρωση σε σχέση με τις αρχικές ε, συνεισφορές των κρατών μελών. Στο τέλος του έτους, ε, ως ηθίστε, θα έχω έχουμε πιστώσεις πληρωμών που θα πρέπει να περάσουν στην επόμενη χρήση. Το ζήτημα είναι να γνωρίζουμε το μέγεθος αυτών των ποσών Αρχικά το 5 με 6 δις, ε, πέρσι φτάσαμε στα 15-16 δις πού θα βρίσκονται αυτά τα αριθμητικά στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να το ξέρουμε και εν πάση περιπτώσει χρειαζόμαστε στοιχεία από, τους, από τις εθνικές διοικήσεις. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς αυτό το ζήτημα και κάθε εβδομάδα θα σας προβάλλουμε πινακοποιήσεις με την εξέλιξη των πληρωμών καθώς και πληροφορίες ως προς τις προοπτικές. Αυτά ήθελα να σας πω σε αυτό το στάδιο των εργασιών για τα πόσα που πρέπει να καταβληθούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αυτός ο τριμερής διάλογος για τις πληρωμές για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Η Μόνικα Χολμάιερ έχει το λόγο. Θα ήθελα... σε σχέση με το κομμάτι του προπολογισμού με τα οποία ασχολούμαι εγώ θα ήθελα από τον Γενικό Διευθυντή να μάθω ποια θα είναι η διαδικασία γιατί βεβαίω θα γίνουν διαπραγματεύσεις, θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Ο Γενικός εισαγγελέα ε, έκανε τις προτάσεις του. Ε, είναι πιθανό το δικαστήριο το Δεκέμβρη να πει ότι κερδι... νικητής θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το Συμβούλιο. Είπανε πολύ κομψά ότι ε, θα ήθελαν κάποια πράγματα να γίνουν ακόμη το 2013. Τι θα γίνει το 2013. Θα υπάρχει ε, καινούριο διορθωτικός προϋπολογισμός. Όλα τα όργανα της κοινότητας θα αλλάξουν τα νούμερά τους. Θα γίνει μεγάλη αναδιάρθρωση. Τι θα γίνει. Θα δεν μπορούν θα αυξήσεις θα κάνουν όλα τα όργανα και μετά θα ξέρουμε ότι θα πρέπει να πληρώσουμε τις αυξήσεις αυτές πότε το 14 αν είμαστε τυχεροί δεν θα γίνει απόφαση, δεν θα πάρθει απόφαση το Δεκέμβριο του 2013, θα πάρθει το 2014 και έτσι θα έχουμε περιθώριο να πληρώσουμε αργότερα. Αν βέβαια η σοφία του Συμβουλίου δεν πάει τόσο μακριά που όσον αφορά τη, το τι ζητούν από τα διάφορα κράτη-μέλη. Αν τώρα ε, το, κοινοβού, το Συμβούλιο λοιπόν ε, υιοθετήσει άλλη στάση δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Ξέρουμε πολύ καλά όμως ότι είναι πολύ πιθανό το Συμβούλιο να ζητήσει ζητήσει να ανακατανεμηθούν κάποια κονδύλια. Γι' αυτό ρωτώ λοιπόν τι θα ζητήσει η Κομισιόν να γίνει τι θα μπορούσε να συμφωνήσει να μην γίνει καμιά αλλαγή ας πούμε ούτε καν στο 13 να πάνε όλα στο 14 εγώ νομίζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι υπερβολικά τεράστιο το έργο που θα πρέπει να κάνουμε το 14. Από εκεί και πέρα θα ήταν πραγματικά δύσκολο και σε, μετά 45 αυτά ε, εκατομμύρια τι θα κάνουμε απλώς θα τα ανακατανύμουμε το 14 το 13 πρέπει να γίνει κάτι για να μην μας πέσουν όλα στο κεφάλι πρόεδρος γενικός διευθυντής πρόεδρε πρώτα πρώτα για τον προπολογισμό του 14 για να απαντήσω στην κυρία Χολμάιερ τον, συντα... τον καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό αυτό βάζοντας τις διοικητικές δαπάνες τα αποτελέσματα μιας ενδεχόμενης θετικής απόφασης για το 11 και το 12 του δικαστηρίου για το 11 και το 12 εμείς η Κομισιόν τώρα το Συμβουλίο για τους δικούς του λόγους αποφάσισε να περικόψει τα ποσά αυτά Άρα αυτό είναι ένα θέμα που θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Προφανώς ο Γενικός Εισαγγελέας έκανε τις προτάσεις του και αυτό δίνει ένα επιχείρημα στο Κοινοβούλιο να ζητήσει την ανασύσταση των σκονδυλίων που περικόπηκαν. Τώρα για το 2013 στο μέτρο που η απόφαση του δικαστηρίου του, μόλις μάλλον πάρθει η απόφαση του δικαστηρίου για το 11 κάθε όργανο θα πρέπει να δει τι ταμείο έχει αν δεν σας ενοχλεί η έκφραση αυτή να το πω έτσι απλά τι έχει στο ταμείο οπότε κάτι θα βρεθεί ακόμη από τις διοικητικές δαπάνες σίγουρα θα στον προπολογισμό του 13 θα υπάρχουν κάποιοι πόροι που δεν θα έχουν ε, απορροφηθεί οπότε θα γίνει μια εκτίμηση θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις στο τέλος του 13 ε, υπάρχει βεβαίως και αύξηση των μισθών ε, αλλά υπάρχει το πάγωμα το αναδρομικό από τον Ιούλιο οπότε δεν θα δοθούν οι αυξήσει των μισθών θα υπάρχουν λοιπόν χρήματα και από εκεί και έτσι θα υπάρχουν κάποια ποσά στα διάφορα ταμεία για να ε, μπαλωθούν κάποια πράγματα Θα δουν λοιπόν τα διάφορα όργανα αν υπάρχουν υπόλοιπα στο 5 και αν όχι τότε θα πρέπει να βρουν άλλες πηγές χρηματοδότησης το οποίο θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα γιατί αφού ο διορθωτικός προϋπολογισμός 2 και ο 8 θα φάνε θα απορροφήσουν όλες τις δαπάνες πληρωμών όλα τις πιστώσεις πληρωμών μέχρι το ανώτατο όριο από πού θα βρεθούν επιπλέον χρήματα μέσω ευελιξίας Τέλος πάντων θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η κατάσταση και από τεχνικής ε, απόψης αλλά και από άποψη χρόνου γιατί αν έρθει αργά η απόφαση του δικαστηρίου τότε θα είναι ίσως να είναι πολύ αργά για την υποβολή ακόμη ενός διορθωτικού προϋπολογισμού. Βεβαίως δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας για το, την, το τμήμα 5. Κυρία Χολμάιερ, θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας αργότερα λοιπόν, μετά το, το, το που θα πάρθει και η απόφαση του δικαστηρίου και αφού θα ξέρουμε τι έχει παραμείνει στα ταμεία των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα διαθέσιμα. Πρόεδρος, ευχαριστώ το Γενικό Διευθυντή. Καλό ήταν να μας δώσετε αυτές τις διευκρινήσεις. Διότι αν ε, βρεθούμε σε μια κατάσταση κατά την οποία ο, ο μόνος ο τρόπος να πληρώσουμε τους μισθούς του προσωπικού θα ήταν μέσω του μέσου ευελιξίας καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι απίστευτα δύσκολα αδιανόητα θα δούμε τις επόμενες μέρες εάν φεύγει καλό ταξίδι στο Βιλνεούς εντωμεταξύ έμαθα και το λέω για τα μέλη του προσωπικού που ε, πρόκειται να πάνε στο στο Βίλνεους απόψε το βράδυ με την Estonian Airlines δεν υπάρχει πια η Estonian Airlines ούτε η πτήση υπάρχει λοιπόν <laughs> κοιτάξτε τι θα κάνετε Λοιπόν, Τώρα πάμε στο θέμα 2 της 4 της ημερήσιας διάταξης πρόκειται για μια μελέτη την οποία έκανε η Deloitte για το εισόδημα των δύο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν κάνω λάθος. Υπεύθυνοι είναι ο Ε, χαιρετώ μάλλον τους, αυτούς που θα μας κάνουν την παρουσίαση και τους συνεργάτες του. Κύριοι, έχετε τον λόγο. Ναι, δέκα λεπτά μας έχουν δώσει για να σας κάνουμε μια παρουσίαση σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής ε, για τα εισόδημα των πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε. Η μελέτη έχει να κάνει με δύο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, ο ο έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όλο το εισόδημα προέρχεται από τέλη που επιβάλλονται στους χρήστες και έτσι δεν υπάρχει ε, συμμετοχή από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και έτσι εξαιρούνται από την απαλλαγή του προϋπολογισμού που χορηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Η μελέτη καλύπτει τον ορισμό των τελών των οργανισμών αυτών, πώς τελικά συλλέγουν τα απαραίτητα κονδύλια. Και κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά την διαδικασία χορηγής επιλογής. Να ξεκινήσω με τα δύο πρώτα σημεία, τον καθορισμό των τελών και τα πλεονάσματα και πώς τα δαπανούν. Κάποια στοιχεία τώρα σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τους οργανισμούς αυτούς, τα τέλεια αυτά θα πρέπει να είναι σε επίπεδα προκειμένου να ισοσταθμίζεται ο προπολογισμό τους. Άρα έξοδα και έσοδα θα πρέπει να ισοσταθμίζονται. Αυτό τι σημαίνει κατά συνέπεια ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ελλείμματα ούτε πλεονάσματα στον προπολογισμό των οργανισμών αυτών. Πώς ε, καθορίζεται λοιπόν το επίπεδο των ελαιών μέσω της επιτροπολογίας. Μας μιλούν και τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί του παρόντος πρέπει να σας πούμε ότι δεν υπάρχουν νομικές προδιαγραφές στο βασικό κανονισμό που να αφορούν ενδεχόμενη παρουσίαση πλανασμάτων εξετάζουμε στη συνέχεια ενδεχόμενα θέματα. Και ο CPVO και ο, OHIM παρουσιάζουν κάποια σημαντικά αποθέματα τα τελευταία χρόνια για τον OHIM 500 εκατομμύρια για τον CPVO 50 εκατομμύρια αυτό τι σημαίνει ότι ο OHIM έχει ε, αρκετά χρήματα για του τριών ετών ενώ ω θα μπορούσε να λειτουργήσει για περίοδο ενό έτου. Άρα θα θεωρούσε κανείς ότι η προδιαγραφή του κανονισμού για τη μην ύπαρξη πλανασμάτων δεν έχει τηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Και πώς καθορίζονται λοιπόν τα τέλη αυτά. Στην παρούσα φάση τα κράτη-μέλη καθορίζουν σε σημαντικό ποσοστό τα τέλη αυτά, το επίπεδο αυτό ενδεχομένως να υπάρχει και ένας κίνδυνος να μην λαμβάνουν υπόψη πάντα υπόψη τα συμφέροντα της Ευρώπης, αλλά βασικά τα συμφέροντα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν σαφείς ε, κανόνες για το τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση ανάκυψης πλεονασμάτων. Δεν είναι εύκολη η για όλα αυτά τα θέματα. Να περάσουμε σε κάποιες από τις αρχές που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές προπτικές των αυτοχρηματοδοτούμενων αυτών οργανισμών σε τήσια βάση, ενδεχομένως να αλλάξει ο τρόπος επιβολής τέτοιων τελών εισφορών, να αλλάξει η διαδικασία της επιτροπολογίας, να καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει και τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε και πιο ακριβείς κανόνες για τον καθορισμό των τελών και συγκεκριμένες προδιαγραφές για το τι θα συμβεί σε περίπτωση συσσόρευσης πλεονασμάτων και πώς θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο στα τέλη προκειμένου ναι, με, ε, να μην υπάρχουν πλεονάσματα αλλά ούτε και ελλείμματα. Έτσι τα τέλη και ο σχετικό ε, κανονισμό θα μπορούσε αυτόματα να τεθεί σε εφαρμογή σε περίπτωση νέα εμφάνιση πλεονασμάτων. Ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε και κάποιες από τις διοικητικέ δομές των οργανισμών προκειμένου να εκπροσωπούν καλύτερα το ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι απαραίτητα τα εθνικά συμφέροντα τόσο πολύ. Και αυτά είναι τα, κάποια από τα βασικά ζητήματα σε ό,τι αφορά ε, τα τέλη και τα πλεονάσματα. Το τρίτο θέμα, το θέμα των, ε, της απαλλαγής για τους πλήρως αυτομοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς έξερονται από την σχετική διαδικασία χορήγησης ε, προϋπολογισμού, απαλλαγής προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012. Έγινε διαθεσμική συμφωνία μεταξύ Επιτροπή Συμβουλίου Κοινοβουλίου, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας λύσης, προβλέπει η υποβολή εκθέσεων από πλευράς των οργανισμών, προκειμένου να υπάρχει πιο πολύ διαφάνεια για τα τέλη, για τα πλεονάσματα και στη συνέχεια ενδεχομένω να υπάρξουν αιτήσει και συστάσεις, αιτήματα και συστάσεις από πλευράς Επιτροπής και Κοινοβουλίου είναι Η δικασία αυτή ενδεχομένως λοιπόν να λάβει η χώρα και να αξιολογηθεί στη συνέχεια για να καθοριστεί κατά πόσο χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα ή όχι. Και έτσι λοιπόν ε, ολοκλήρωσα την σύντομη αυτή παρουσίασή μου σε ό,τι αφορά τα βαστικά σημεία που περιλαμβάνει η μελέτη αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σαφέστατη παρουσίαση. Οκ. Οκ. Οκ. Euh, λοιπόν, η συγγήτρια. Θέλετε και μετά η Ούτε Χάουκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, νομίζω ότι η μελέτη καταδεικνύει με σαφήνεια ότι εδώ συμβαίνουν πράγματα ιδιαίτερα εν ώψη της οικονομικής κρίσης, τα οποία δεν είναι απαραίτητα επιθυμητά. Βάσει λοιπόν της ε, βάσης αυτής ε, και βάσει της, ε, των κανονισμού, αν δεν επιτρέπεται η συσσωρευσή πλεονασμάτων, παρόλα αυτά αυτό συμβαίνει, το θέμα που ανακύπτει είναι τι κάνουν τα κρατημέλη. Και αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερως είναι το εξή. Από ό,τι φαίνεται, από χρονικής άποψη δεν ε, μπορούμε να προβλέψουμε τέτοια πρόστιμα σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς. Δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως στο έπακρον. Και εμένα αυτό που με καταδεικνύει αυτή η μελέτη είναι ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει πολιτικός διάλογος για το πώς θέλουμε να διαρθρώσουμε, να δομήσουμε καλύτερα την κατάσταση αυτή. Ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε από τη μελέτη αυτή, πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε διαφορετικά και άλλους οργανισμούς. Το θέμα δεν είναι να κόψουμε τα φτερά και τον προπολογισμό των ε, ε, οργανισμών αυτών μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν πλεονάσματα, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι ε, θα διαβάσω την μελέτη. Πολλά καλά σημεία μας κατέδειξε και η παρουσίαση. Το σημαντικό είναι να το σκεφτούμε από τώρα. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε και τι μπορούμε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμβάλλουμε για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής. Γιατί άλλο να υπάρχει κάποια ισορροπία στον προπολογισμό από την δημιουργία πλενάσματων και ελλημάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, παράδεικτο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά σε, ό,τι σχέση και με την οικονομική κρίση. Πραγματικά είναι πνευματικό. Ευχαριστώ, η Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η μελέτη αυτή πραγματικά είναι πολύ ωφέλιμη. Ειλικρινά. Μεταξύ άλλων, επειδή επιβεβαιώνει και την προσέγγιση τη δική μας. Ό,τι λέμε δηλαδή ότι και οι δύο οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Και οι δύο οργανισμοί έχουν ως εκ δικαίωμα να ζητούν τέλη, εισφορές από τις επιχειρήσεις. Αλλά θα πρέπει οι εισφορές αυτές από τις επιχειρήσεις να είναι μόνο τόσες ώστε να, χρειά... να αυτό χρηματοδοτούνται. Όχι σε παραπάνω ε, εισφορές. Η ιδέα την οποία γέννησε το Συμβούλιο το 2010 ήταν η εξή. Οι οργανισμοί τα πλεονάσματα αυτά να τα μεταφέρουν στις εθνικές υπηρεσίες, στην εθνική κυβέρνηση. Βρήκαν και κάποια, κάποιους τύπους για την κατανομή των πλεονασμάτων αυτών. Αυτό δεν απο... θεωρώ ότι είναι ανοησία, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Γιατί, επαναλαμβάνω ότι οι υπηρεσίες, οι οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες για επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να αποτελούν μέσο έμεσης ε, φορολόγησης για τις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι παράλογο και δεν αποτελούν το σκοπό μας. Γι' αυτό θεωρώ λοιπόν ότι οι προτάσεις που καταβάλλονται για το πώς θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, τροποποιήσεις, πώς ενδεχομένως να βρούμε ένα επίπεδο αυτόματο, αυτόματο υπολογισμού των εισφορών, το οποίο ενδεχομένως να αυξάνεται όταν δεν επαρκούν οι εισφορές αυτές σε περίοδο δύο ετών ή να μειώνεται αντίστοιχα βάσει διαφορετικής ε, δομής των εισφορών. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό αποτελεί μια πολύ καλή ιδέα. Και σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί σε πολλές ε, περιπτώσεις δεν μιλάμε για την ε, ιατρική, για τη χημική βιομηχανία. Υπάρχουν άλλες εισφορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως να μην προβλέψουμε να μην υπάρχουν και καθόλου εισφορέ για αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, ίσως λόγω λανθασμένων ε, υπολογισμών να επιβλήθηκαν λανθασμένε εισφορές. Αυτό θεωρούσε ότι θα ήταν μια καλή λύση, όχι όμως με Τέτοια ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκές εισφορές τελικά να χρηματοδοτούνται οι εθνικές κυβερνήσεις, οι εθνικές διοικήσεις. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την πραγματικά πάρα πολύ καλή σύνοψη και για την πολύ καλή μελέτη. Ε, merci Jutta, Monika Also möchte Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω πραγματικά τη Γιούτα Ποιος σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να προβλέπεται δυνατότητα μέσω εισφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο να χρηματοδοτούνται εθνικά, εθνικές υπηρεσίες, η εθνική διοίκηση. Να υπάρχει τέτοια επιδότηση, τι να πω, πιστεύω ότι είναι πραγματικά μεγάλη ανοησία και πραγματικά μας μπλέκει και αυτή η αδιαφάνεια που υπάρχει, αυτή η, η των πόρων σε ό,τι αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πω ότι οι εισφορές έχουν αυξηθεί και αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις αυτές. Και αντιμετωπίζουμε παράλληλα μια κατάσταση όπου οι οργανισμοί δεν μπορούν να έχουν το επαρκές προσωπικό για να ανταποκρίνονται στα αιτήματα, τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που έχουν. Γι' αυτό λοιπόν να πω ότι στην παρούσα φάση έχω την αίσθηση ότι δεν είναι λογική η αντιμετώπιση, είναι μάλλον συναισθηματική. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια καλύτερη λογική ανάλυση. Σας ευχαριστώ και για τη μελέτη. Θεωρώ ότι κατά πρώτον θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, αυξάνονται υπερβολικά οι εισφορές, να μην επιβαρύνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης όταν τελικά συλλέγονται αυτοί οι πόροι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ίδιο το προσωπικό των οργανισμών. Ίσως ε, και σε ό,τι αφορά τις νέες εντολές, ε, τις ε, νέες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν, να πρέπει να υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση. Όταν ξαφνικά, για παράδειγμα, ένα οργανισμό λαμβάνει 6.000 δείγματα παραπάνω, χρειάζεται και τον έργο προσωπικό για να τα διεκπαιρεώσει. Όλα αυτά που συζητάμε λοιπόν εδώ έχουν ε, σημαντικό αντίκτυπο και θα ήθελα να υποστηρίξω λοιπόν την θέση της Γιούτα Χάουγκ. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις. Θέλετε να σχολιάσετε για όσα προελέχθησαν. Τα σχόλια που άκουσα συμβαδίζουν με τις συστάσεις της μελέτης και ελπίζω να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στην πορεία σας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη. Όπως είπαν και οι παρεμβαίνοντες και οι συγγήτρια, βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση όπου υπάρχουν πλεονάσματα με τα οποία δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και ένα θέμα διαχείρισης. Ευχαριστούμε για την ανάλυση και τις συστάσεις που είναι χρήσιμες για την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ πολύ και σας απελευθερώνω, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας προτείνω να σταματήσουμε τις εργασίες μας, να διακόψουμε τις εργασίες. Είχαμε προβλέψει ψηφοφορία το απόγευμα στις 3. Προτείνω να ψηφίσουμε τώρα. Αλλά επειδή δεν έχω τους υπευθύνους εδώ να με πλαισιώσουν, έχουμε και άλλους προσκεκλημένους που έρχονται και θα παρευρεθούν στην αναστολή της συνεδρίασης στη διακοπή της συνεδρίασης. Euh, Από σένα προέρχονται, δικοί σου προσκεκλημένοι είναι. <laughs> Δεν μπορούμε καν να τους πούμε ότι κάνουμε διακοπή γιατί δεν φορούμε τα ακουστικά τους. it's a, a bus full of yeah, uh, bus, visitors yeah. and. Uh... Je salue les les visiteurs. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους προσκεκλισμένους. Μα, με ακούτε; Α, με ακούν οι προσκεκλημένοι του Ράιμαρ Πέγγ από το Σλέσφιγ Χολστάιν. Σας ε, χαιρετίζω, σας καλωσορίζω, αλλά φτάνετε μία στιγμή όπου διακόπτουμε τις εργασίες μας. Μπορείτε να συνεχίσετε εσείς. Αλλά έληξαν οι πρωινές μας εργασίες ή το σημαντικό το θέμα. Μιλήσαμε για το σχέδιο προϋπολογισμού του 14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς ε, χρηματοδοτείται, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, ποια είναι η χρησιμότητά του. Άλλοι φίλοι σας συμμετείχαν νωρίτερα σε εργασίες μας, έχουν λήξει όμως οι εργασίες και διακόπτουμε μέχρι τις 3 το απόγευμα και θα αρχίσουμε στις 3 με ψηφοφορίες. Σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μας θυμάται, αλλά λυπούμεθα που δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε μια πραγματική συζήτηση Επιτροπής Προϋπολογισμών. Λοιπόν, διακόπτεται η συνεδρίαση, θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα.